ένταση στη Μέση Ανατολή. Είμαι από τη Βουλγαρία και είμαστε στην πρώτη γραμμή ε, της συρροής των μεταναστών και προσφύγων και σίγουρα η έξαρση των εντάσσεων στη Μέση Ανατολή δημιουργεί νέες απειλές. Επίσης, ε, θα πρέπει να γίνει μετακατάσταση περίπου 2 εκατομμυρίων ε, προσφύγων στις κουρδικές περιοχές ε, λόγω των επιχειρήσεων του τουρκικού στρατού. Κατά τη γνώμη μου, η μετακατάσταση θα πρέπει μόνο οικειοθελώ να γίνει και όχι η βάρο του τοπικού κουρδικού πληθυσμού. Μία αλλαγή του εθνοτικού, της εθνοτικής κατανομής ε, και του χάρτη των εθνοτήτων θα δημιουργήσει μία μόνιμη απειλή για μεταναστευτικές ροές από τις κουρδικές περιοχές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό καλό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προτείνει ένα διεθνή μηχανισμό για τη διαφάνεια και τον έλεγχο αυτών των μεταναστευτικών ροών. κυρία Χέινα για ένα λεπτό. Ο κύριος, συγγνώμη, Χέινα Κύριε Πρόεδρε, ναι βεβαίως όλοι λυπούμεθα για αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή καθημερινά. Πεθαίνουν άνθρωποι στη Συρία, στο Ιράν, τα ανθρώπινα δικαιώματα παραβιάζονται, ακόμα και στο Ιράκ εκ νέου προκύπτουν προβλήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. και βεβαίως ε, παραβίωση τα δικαιώματα των ανθρώπων που διαδηλώνουν. Όλα αυτά συμβαίνουν αφότου οι Αμερικανοί και οι σύμμαχοί τους ε, εισέβαλαν στο Ιράκ και αυτό δημιούργησε μεγάλη ανισορροπία στην ευρύτερη περιοχή. Οδήγησε σε ανεξέλεγκτη βία που δεν έχει σταματήσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι σαφή σε αυτά που λέει, πρέπει να υποστηρίξει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία όμως ε, χρειαζόμαστε ε, οπωσδήποτε υπομονή, διότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται εύκολα και απλά. Ευχαριστώ κύριο Τσουχοντάρου για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Βηρητός, ε, Βαγδάτη, Τεχεράνη, ε, τρεις, τρία σημεία καυτά αυτή τη στιγμή. Αντί για ψωμί και δημοκρατία, ο κόσμος ε, ε αντιμετωπίζεται με βία πολλοί φίλοι μου, γιατροί εκεί, συνάδελφοί μου ενώ πεθαίνουν εκεί προσπαθώντας να γιατρέψουν, να, να, να ασχοληθούν με τους τραυματίες. Ε, χρειάζεται ε, προστασία, χρειάζεται διαφάνεια για αυτά που συμβαίνουν εκεί. Θέλω να πω στην είπατε εκπρόσωπο τι μέτρα αφήνετε για, την, για το διάδοχό σας για να μην συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και υπάρχει κάποιο ε, χρονοδιάγραμμα, κάποια προθεσμία για να εφαρμοστούν αυτά. Σας ευχαριστώ. Στη διαδικασία του Catch the Eye έχω λάβει εξαιτήματα. Να υπενθυμίσω ότι οι ομιλητές έχουν στη διάθεσή τους ένα λεπτό καθένας. Πρώτο κύριο κύριος Γιζίπος Σπίσελ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, κυρία Μογκερίνη για την ε, δουλειά που έκανε σε ολόκληρη αυτήν την θητεία. Δεν συμφωνούσαμε πάντα. Εγώ θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ θετική απέναντι στο καθεστώς ε, του Ιράν και πολύ αισιόδοξη και τώρα φαίνεται ότι έχει φτάσει η στιγμή ε, να αξιολογήσουμε πώς θα έπρεπε να είμαστε πιο σκληροί. Οι κοινωνικές συνθήκες είναι συγκλονιστικές. Έχουμε τεράστια διαφθορά σε κάθε πόλη είναι κάπως διαφορετικό το καθεστώς. Αλλά είναι αναγκαίο η Κομισιό να αξιολογήσει μήπως ε, θα πρέπει να είμαστε κάπως πιο ε, αυστηροί απέναντι στο Ιράν γιατί αποτελεί μια πηγή αποσταθεροποίησης στη Μέση Ανατολή και καταπίεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πρέπει να φροντίσουμε βεβαίω να μην εκμεταλλευτούν την ευκαιρία αυτή οι Ισλαμιστές. Ο κύριο Χουάν Φερνάντο Λόπε Αγγιλάρ. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Αντιπρόεδρε, Σήμερα, με μεγάλη πλειοψηφία, εγκρίναμε την Επιτροπή τη κυρία Φοντερ Λάινεν. Θα ήθελα και εγώ να αναγνωρίσω και να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για το σκληρό έργο σα και τι εργόδε σα προσπάθειε την τελευταία πενταετία και πραγματικά μέχρι αργά το βράδυ να κάθεσαι εδώ για να συζητούμε την κατάσταση σε τρει χώρε της Μέση Ανατολή που δεν έχουν και πολλά κοινά σημεία μαζί του. Το πιο κοινό του σημείο είναι οι διαδηλώσεις και η αστάθεια. Ο Λίβανος ε, Την αστάθειά του την οφείλει στην ανάμειξη του Ιράν τα τελευταία χρόνια. Και μεταξύ του Ιράκ και του Ιράν είχαμε έναν ε, ματηρό πόλεμο. Βέβαια, η πιο ανησυχητική κατάσταση είναι αυτή του Ιράν, γιατί αυτή είναι εκείνη που κρατάει περισσότερο και μάλιστα είχαμε κλιμάκωση το, της καταπίεσης, ιδιαίτερης βάρος των γυναικών. Και έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό εκτέλεση θανατικών ποινών εκεί. Και επίσης ε, έχουμε πολλούς ε, νεκρούς και πάρα πολλούς τραυματίες. Έχουμε και την Ήτα μία, ένα κορίτσι 14 ετών και μάλιστα η χρήση της βίας όχι μόνο είναι δυσανάλογη από το Ιράν, αλλά και συστηματική για να γίνει βάναυση κατά πίεση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας. Φυσικά συμφωνούμε με την Πυρηνική Συμφωνία, αλλά δεν μπορούμε να σιωπούμε μπροστά σε αυτή τη συστηματική βαναυσότητα του Ιρανικού καθεστώτος. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Ανθία Μακιντάιερ για ένα λεπτό επίσης. We really just δεν μπορούμε να καθόμαστε και να αγνοούμε αυτά που συμβαίνουν στο Ιράν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η διεθνής κοινότητα πρέπει οπωσδήποτε να καταγγείλουν την ε, μαζική χρήση βίας από την ε, ε, φρουρά την Ιρανική, από το Ιρανικό καθεστώς. Ο θάνατος 143 ανθρώπων έχει καταγραφεί από την Διεθνή Αμνηστία. Όμως ε, θεωρούν ότι ο αριθμός των νεκρών είναι υψηλότερος και οι περισσότεροι από τους νεκρούς έχουν πυροβοληθεί, όπως ο Νίκταρ Ισταντάνη. Ήταν 14 χρονών και πυροβολήθηκε στο κεφάλι. Η οικογένειά της την έψαχνε για τρεις μέρες, έως ότου της δώσουν τη σωρό ε, το καθεστώς η απάντησή μας έως τώρα δεν ήταν η κατάλληλη. Πρέπει να ζητήσουμε από τους ηγέτες αυτού του καθεστώτος να δρογοδοτήσουν για τα εγκλήματά τους. Δεν μπορεί να υπάρξει κοινή επιτροπή με το Ιράν όσο το καθεστώς του Ιράν προβαίνει σε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Κλέρ Ντάλι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και χάρηκα ιδιαίτερα που η κυρία Μογκερίνη μίλησε για το ότι η Ευρώπη είναι αντίθετη με την μονομερή αποχώρηση τον ΗΠΑ από την ε, Συμφωνία για τα Πυρηνικά του Ιράν. Αλλά πρέπει να πάμε παραπέρα και να αναγνωρίσουμε ότι οι κυρώσεις κατά του Ιράν έχουν προκαλέσει μεγάλες δυσκολίες στους πολίτες ε, του Ιράν, ειδικά στους ανθρώπους που λέμε ότι πρέπει να προστατεύσουμε. Και τώρα έχουμε το εξή θέαμα. Οι ΙΠΑ προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τις θεμητές ε, και αυθεντικές διαμαρτυρίες ε, στο Ιράν και στον Λίβανο για να χτυπήσουν το Ιράν. Δεν πρέπει να πέσουμε στην παγίδα. Ο Μάικ Πομπέο λέει ότι αυτά προκαλούνται από την διαφθορά. Είναι πραγματικοί άνθρωποι με πραγματικά προβλήματα. Η διαφθορά, η πανάπτυξη, μια καταστραμμένη οικονομία, τα αποτελέσματα του πολέμου με το Ιράκ. Δεν πρέπει να πέσουμε στην παγίδα των ΗΠΑ πρέπει να εργαστούμε για την σταθερότητα στις ε, χώρες αυτές και για ειρήνη στην Ιεμένη. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Μικ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ κυρία Μογκερίνη θεωρώ ότι στην εισφορά σας ε, για το Ιράν ε, είναι πολύ πιο ισορροπημένη από αυτά που είπαν άλλοι οι εξελίξεις στο Ιράν, στο Ιράκ και στο Λίβανο είναι διαφορετικές μεταξύ τους. Έχουν... Αλλά υπάρχει και κάτι κοινό. Ε, όλοι έχουν υποφέρει από διεθνείς, διεθνείς συνεχείς διεθνείς παραμβάσεις, ε, εμφύλιους πολέμους, διεθνείς κυρώσεις ε, και βεβαίως ε, ε, οι φυσικοί πόροι οι οποίοι έχουν λιελατηθεί. Οι άνθρωποι αυτοί που πεθαίνουν στις χώρες αυτές ο κάθε ε, διαδηλωτής ο οποίος ε, σκοτώνεται από, την Ιρανική, από το Ιρανικό καθεστώς πρέπει να το καταγγέλουμε. Βεβαίως κάποιοι χρηματοδοτούν την αντιπολίτευση στο Ιράν για να προσταθεροποιηθεί η κυβέρνηση, διεθνείς δυνάμεις. Πρέπει λοιπόν να καταδικάζουμε τους θανάτους ε, των ε, διαδηλωτών και στο Ιράκ και στο Λίβανο. Πρέπει επίσης να καταδικάζουμε τον θάνατο των διαδοτών στη Βολιβία και στο Ιράν. Ας είμαστε δίκαιοι. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μάρτιν Πάτεν έχει το λόγο για ένα λεπτό. Λυπούμε για τους ε, θανάτους ε, και τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν και την κράτηση πολιτικών ε, κρατουμένων που πρέπει να απελευθερωθούν αμέσως. Αλλά η πρώτη προτεραιότητα στο Ιράν είναι να μην φτιάξει πυρηνικά όπλα. Αλλά τώρα ξεκινάει ξανά τον εμπλωτισμό του ουρανίου. Στηρίζω λοιπόν την ε, σχετική συμφωνία, αλλά πρέπει να προετοιμαστούμε για την αποτυχία της και να αναζητήσουμε ένα εναλλακτικό σχέδιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αθώα για αυτό το χάλι. Το σχέδιό της για την παράκαμψη των κυρώσεων του ΟΗΕ τώρα κατέληξε στο να απειλείται η Ευρωπαϊκή Ένωση με αντίπεινα. Θα πρέπει λοιπόν να βρεθεί μια λύση με την ενεργό συμμετοχή των ΙΠΑ. Ε, Πολλοί εδώ πέρα καταγγέλουν τον πρόεδρο Τραμπ, αλλά αν θέλουμε η Μέση Ανατολή να μείνει χωρίς πυρηνικά και αν στηρίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ιρανών, πρέπει να αποκαταστήσουμε τις φιλίες μας με την Ουάσιγκτον, όχι την Τεχεράνη. Είμαι σίγουρο πω η σχέση τη Βρετανία με τις ΙΠΑ θα βοηθήσει. Σας ευχαριστώ και τώρα το λόγο έχει η Αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η εκπρόσωπο για τι εξωτερικέ σχέσει, η κυρία Φεντερίκα Μογκερίνη. Σα ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Διαπιστώνω ότι η πλειοψηφία των Ευρωβουλευτών ε, επιβεβαίωσε και ενθάρρυνε την προσέγγισή μας, αυτή που σας περιέγραψα κατά την έναρξη της συζήτησης. Και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Θα ήθελα να απαντήσω σε μία ερώτηση που τέθηκε από κάποιον που στο μεταξύ έφυγε, ε, από μία ευρωβουλευτή μάλλον που έφυγε. Είμαι σίγουρη ότι μας παρακολουθεί με προσοχή από το γραφείο της. Ε, απευθύνει έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να χρηματοδοτήσει ειδικά προγράμματα στη Μέση Ανατολή και ανέφερε ιδιαίτερα τη θέση του Ιράκ. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να σας δώσω κάποια στοιχεία. Για το Ιράκ μόνο, έχουμε χρηματοδοτήσει συγκεκριμένα σχέδια και προγράμματα για την αποναρκοθέτηση, τη δημιουργία θέσεων απασχόληση, την επανασυμφιλίωση. Σχέδια που υπάρχουν, που επισκεφτόμαστε και ελέγχουμε συνεχώ Και εγώ προσωπικά και η αντιπροσωπεία μας επιτόπου. Και φαντάζομαι και εσεί τα έχετε επισκεφθεί. Μερικά προγράμματα από αυτά που χρηματοδοτούμε στη Μέση Ανατολή. Για το Ιράκ τα τελευταία χρόνια 1,25 δισεκατομμύρια ευρώ έχουμε αφιερώσει σε συγκεκριμένα σχέδια μόνο για το Ιράκ. Και δεν περιοριζόμαστε όπως βλέπετε μόνο στη διπλωματία. Παρόλο που η διπλωματία στους καιρούς αυτούς και με τη διεθνή πολιτική κατάσταση, η διπλωματία σίγουρα είναι ένα πολύτιμο στοιχείο και μερικές φορές ε, υποτιμούμε, πιστεύω, την ε, ισχύ της διπλωματικής μας ε, ανάμειξη και δέσμευση. Αλλά δεν περιοριζόμαστε μόνο στη διπλωματία. Στηρίζουμε συγκεκριμένα προγράμματα και σχέδια που βελτιώνουν την καθημερινότητα. Γιατί είπε κάποιο ότι είναι πραγματικοί άνθρωποι, είναι πραγματικέ ανάγκε. Άνδρε και γυναίκε που αντιμετωπίζουν δυσκολίε όχι μόνο χρόνια ολόκληρα, δεκαετίε ολόκληρε. Και διαβιούν σε πολύ αντίξωε συνθήκε και από άποψη οικονομική και από άποψη ασφάλεια. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα θεσμικά τη όργανα χρηματοδοτούμε τέτοια συγκεκριμένα ε, προγράμματα που πραγματικά σώζουν τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων στην περιοχή. Και θα περίμενα να το γνωρίζουν αυτά, αυτό οι ευρωβουλευτές. Οπότε ε, ενημερωθείτε, κατατοπιστείτε τουλάχιστον για τα προγράμματα που έχετε συμφωνήσει και εσείς να χρηματοδοτήσουμε στην περιοχή. Νομίζω αν είστε καλύτερα ενημερωμένοι θα ε, προσωπείτε καλύτερα και τους ψηφοφόρους σας. Επίσης, δεν μπορώ εγώ να προδικάσω την πολιτική και τη θέση του διαδόχου μου, του είπα το εκπροσώπου για την εξωτερική πολιτική, ούτε τη θέση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή με το Συμβούλιο θα διαμορφώσουν την άποψή του. Πάντω, ελπίζω και πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα συνεχίσει στο μέλλον και θα είναι σημαντικός εταίρος και αυτό χάρη του τοπικού πληθυσμού, γιατί μερικές φορές δεν αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος μας. Κάθε φορά που επισκεφτόμαστε την περιοχή, ακούμε από τους συνομιλητές μας, από τον απλό κόσμο, την κοινωνία των πολιτών, όχι μόνο από τους ε, κυβερνώντες και τους ε, φορείς, τους θεσμικούς. Όλοι αναγνωρίζουν το ρόλο μας. Πολύ περισσότερο από ότι οι Ευρωπαίοι μερικές φορές. Οπότε θα πρέπει να συνεχίσουμε τις επενδύσεις και να τις ε, ενισχύσουμε σε οικονομικό επίπεδο, σε επίπεδο διπλωματίας, αλλά και ε, στην ασφάλεια και να στηρίξουμε αυτή την περιοχή για να βρει το δρόμο της προς βιώσιμη ειρήνη και ασφάλεια. Και όπως είπαμε ε, και στην αρχή, θα πρέπει να στυλιτεύσουμε αμήλικτα οποιαδήποτε μορφή βίας και ιδιαίτερα ε, την καταπίεση των διαδηλωτών με δυσανάλογη χρήση βίας από τις αρμόδιες αρχές. Και στο Ιράκ επίσης έχουμε ε, εμπλακεί και στον τομέα της ασφάλειας, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει ανάγκη μεταρρύθμισης αυτού του τομέα. Και θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας, γιατί διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ανάγκη αλλαγής και βελτίωσης του τρόπου λειτουργίας ε, των θεσμών, των φορέων ασφάλειας ε, της χώρας. Οπότε, επαναλαμβάνω και πάλι την ελπίδα μου ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα στηρίξει αμέριστα περαιτέρω δέσμευση και προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των θεσμικών της οργάνων στην περιοχή. Θα δώσω τώρα τη σκητάλη στο συνάδελφο Μίμητσα και τα λέμε αύριο πάλι. Μάλιστα, ευχαριστώ κύριε Πατεκπρόσωπε. Ολοκληρώνουμε τη συζήτηση για το θέμα αυτό. Και περνάμε, τώρα στο επόμενο, σημείο της ημερήσιας διάταξης. Τις ενεξελίξει διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών ΑΚΕ. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι μπορείτε να ζητάτε το λόγο με, για τη διαδικασία της υποβολής ερώτησης με μπλε κάρτα και με το συνήθι τρόπο αλλά και ηλεκτρονικά. Θα δώσω τώρα το λόγο στον, ε, στον πρόεδρο της Επιτροπής Ανάπτυξης, τον κύριο Τομπέ, για πέντε λεπτά, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ε, κύριε Επιτροπέ, κυρία Υπουργέ. Ε, σα ευχαριστώ που είστε εδώ τόσο αργά. Η συμφωνία του Κοντονού μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών ΑΚΕ, Αφρικής, Καραβικής, Ειρηνικού, είναι η πιο πλήρης ε, σύμπραξη που έχει συμπράξει ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Συμφωνία του Κοτονού καλύπτει συνεργασία με περίπου 80 χώρες παγκοσμίως... και καλύπτει ένα ευρύ πεδίο τομέων πολιτικής. Είμαστε σε μια εποχή όπου υπάρχει όλο και μεγαλύτερη ανασφάλεια. Εμείς λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υπερασπιστούμε και να προωθήσουμε τον πολυμερή χαρακτήρα, τη διεθνή συνεργασία, και ένα νέα, μια νέα τάξη πραγμάτων που αναβασίζεται σε κανόνες. Αυτή είναι βασικά, βασικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Φεβρουάριο του, 2020 ολοκληρώνεται η Συμφωνία του Κοτονού. Οι διαπραγματεύσεις για τη νέα συμφωνία έχουν ήδη ξεκινήσει. Νωρίτερα το Κοινοβούλιο έχει αναφέρει τι θέλουμε να περιλαμβάνουν αυτή η νέα συμφωνία. Οι ανησυχίες του Κοινοβουλίου ε, θα ληφθούν υπόψη όταν ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση. Ε, έως τώρα έχει υπάρξει συμφωνία ότι η νέα σύμπραξη θα πρέπει να βασιστεί σε βασικές αρχές ε, και αξίες. Ε, με τη συμφωνία αυτή υπάρχουν και τρία περιφερειακά πρωτόκολλα, πρωτόκολλα που θα αναφέρουν τους, τις προδιαγραφές, προδιαγραφές συνεργασίας ανάλογα με την κάθε περιοχή θα πρόκειται για ένα ενιαίο νομικό δεσμευτικό μέσο. Αυτό δεν ήταν προφανές, όμως είναι ένα από τα βασικά, ήταν ένα από, τα βασικά αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στη σημερινή συζήτηση ε, χρειαζόμαστε μεγαλύτερη σαφήνεια και βεβαίως θα χρειαστούμε και, και ένα νέο ψήφισμα, διότι ε, κάποιες από τις βασικές ανησυχίες του Κοινοβουλίου δεν έχουν καλυφθεί. Εκ μέρου τη Επιτροπή Ανάπτυξη έχουμε υποβάλει ερωτήσει προ το Συμβούλιο και προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλουμε να ακούσουμε λοιπόν σαφεί απαντήσει στα ερωτήματα αυτά σήμερα. Θεωρούμε ότι τα ερωτήματα αυτά θα μα δώσουν κατευθυντήριε γραμμέ ε, και εν ώψη τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το πρώτο ερώτημα είναι λοιπόν πού βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά το βασικό αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η νέα συμφωνία να ενισχύσει την ε, κοινοβουλευτική διάσταση σε επίπεδο χωρών ΑΚΕ. Θέλω εδώ να κρατήσω σαφέ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να δεχτεί το εκτελεστικό επίπεδο της εξουσίας να μην έχει κάποιον, ε, κάποιο αντίστοιχο επίπεδο κοινοβουλευτικό. Να έχουμε δηλαδή κοινή επιτροπή ε, ε, μεταξύ εκτελεστικών εξουσιών και να μην υπάρχουν κοινοβουλευτικές ε, συναντήσεις. Εμείς συμφωνούμε με του τρει πυλώνες, όμως αυτό δεν αρκεί, τους τρεις πεζακούς πυλώνες, αλλά δεν αρκεί αυτό. Δεν θέλουμε να χαθούν ε, τα ωφέλη μιας συζήτηση μεταξύ ομοτήμων σε επίπεδο ΑΚΕ. Ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα και εκ μέρου τη επιτροπή μας. Το Συμβούλιο, η Επιτροπή, ε, ποια είναι η άποψή τους όταν μιλάμε για την καταπολέμηση ε, των διακρίσεων λόγω του φύλου, λόγω των σεξουαλικών προτιμήσεων, πώς θα, εξασφαλίσουμε ότι τα αναπορευγικά δικαιώματα θα συμπεριληφθούν σε αυτή τη νέα συμφωνία. Είναι βασικές κεντρικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα ληφθούν υπόψη στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας. Ένα άλλο σημαντικό ερώτημα έχει να κάνει με την κοινωνία των πολιτών. Σε κάποιες χώρες πρόκειται για ένα σοβαρό λόγο ανησυχίας. Θέλουμε να αυξηθεί ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών και για να συμβεί αυτό ε, θα πρέπει να αναφέρεται στη συμφωνία σε όλα τα επίπεδα. Τέλος, το Κοινοβούλιο είπε ότι η νέα συμφωνία πρέπει να προβλέπει ένα νέο μηχανισμό παρακολούθησης της πρόοδου και παρακολούθηση των κενών για την εφαρμογή των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Χρειαζόμαστε λοιπόν μεγαλύτερη σαφήνεια τελικά πώς αυτά θα ενσωματωθούν στην επόμενη συμφωνία. Πριν ολοκληρώσω όμως ε, με ένα σαφές μήνυμα του Κοινοβουλίου θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επίτροπο, τον κύριο Μίμικα για την πολύ σκληρή δουλειά του τα τελευταία πέντε χρόνια. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για αυτή τη συνεργασία έως τώρα ε, και βεβαίως και το Συμβούλιο βασιζόμαστε στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προωθήσουν, να στηρίξουν τα αιτήματά μας στις επόμενες εβδομάδες και μήνες και να μας δώσουν και απαντήσεις σήμερα, σαφείς απαντήσεις κατά προτίμηση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Εκ μέρους του Συμβουλίου τώρα, το λόγο έχει η Υπουργό Τίτη Τουπουράινεν. Παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, Είναι τιμή μου που σας μιλάω σήμερα για τις ε, διαπραγματεύσεις μεταξύ των χωρών ΑΚΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για μια πολύ επικαιρή συζήτηση. Η κατάσταση μετά τον Κοτονού είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για το Συμβούλιο. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Μέχρι στιγμή είχαμε πέντε γύρους διαπραγματεύσεων στο πολιτικό επίπεδο. Τελευταίος τον Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη. Η επόμενη συνεδρίαση των επικεφαλής διαπραγματευτών θα γίνει τον Σεπτέμβριο και τα δύο μέρη συμφωνούν ότι το νέο πλαίσιο θα πρέπει να βασίζεται στην ατζέντα του 2030 και την Συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή και θα πρέπει να προσαρμοστεί στο νέο παγκόσμιο πλαίσιο τις νέες προκλήσεις και ευκαιρίες. Οι φιλοδοξίες είναι ψηλές και από τις δύο πλευρές για να χρησιμοποιήσουμε την σχέση μας για κοινέ θέσει στα διεθνή φόρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνεί με την φιλοδοξία της μεικτής Κοινοβουλευτικής ε, Συνέλευσης ε, ΑΚΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να ενισχύσουμε την ε, σχέση μας. Οι διαπραγματευτικές μας οδηγίες λένε ότι τα μέρη θα έχουν μια ανοιχτή προσέγγιση που θα σκοπεύει να ενισχύσει τον ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων, τοπικών αρχών, της κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα. Οι οδηγίε αυτέ έχουν στόχο να ενισχύσουν τον τακτικό πολιτικό διάλογο σε όλα τα επίπεδα για να υπάρχει η εμπλοκή διαφόρων ενδιαφερομένων της κοινωνίας των πολιτών στις διαδικασίες του διαλόγου. Επίσης έχουν στόχο να ενισχύσουν τον ρόλο της κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα ως βασικών εταίρων στην υλοποίηση των στόχων αυτών. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι βουλευτέ, οι διαπραγματεύσει στα ζητήματα μετανάστευση συνεχίζονται. Στόχο τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να καταλήξουμε σε ένα πιο επιχειρησιακό κείμενο σε σχέση με τη Συμφωνία Κοτονού. Η διαπραγματευτική εντολή επίσης ορίζει ότι όλα τα στοιχεία αυτά θα αναφερθούν στον τακτικό πολιτικό διάλογο, κατά το οποίο σημαίνει ότι θα έχουμε τακτικές συζητήσεις με τους εταίρους μας για αυτό το σημαντικό θέμα. Οι συμφωνίες οικονομικής συνεργασίας βοηθούν τις κοινότητες με το να παρέχουν την απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη την ε, τεχνολογία και την πύρα Είναι λοιπόν εργαλεία τα οποία βοηθούν στην ε, αύξηση της προσθέμενης αξίας, ε, την οικονομική ένταξη και τη βιομηχανοποίηση. Θα πρέπει λοιπόν αυτά να αποτελέσουν υπόδειγμα και για τις μελλοντικές εμπορικές μας σχέσεις. Οι διαπραγματευτικέ οδηγίες της Ένωσης είναι πολύ σαφείς όταν μιλάμε για μη διακριτική μεταχείριση ε, με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Στόχος είναι να δεσμευτούν τα μέρη στην προαγωγή των δικαιωμάτων όλων των ατόμων για να μπορούν να αποφασίζουν ελεύθερα και υπεύθυνα για ζητήματα που αφορούν την σεξουαλικότητά τους και την αναπαραγωγική τους υγεία ε, χωρίς βία και καταναγκασμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στόχο να υπάρξει μια συμφωνία που θα διασφαλίζει καθολική πρόσβαση σε υπηρεσίες ε, υγείας ε, και εκπαίδευσης για τα ζητήματα αυτά περιλαμβανομένης της ε, σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Ευχαριστώ. Εκ μέρους τώρα της Επιτροπής, το λόγο έχει ο Επίτροπος Νέβεν Μίμητσα, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμη Ευρωβουλευτέ, κύριε Υπουργέ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Τομπέ, τον πρόεδρο της Επιτροπής Ανάπτυξης και όλα τα μέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης για το εξαιρετικό τους έργο και για την πολύ στενή συνεργασία που είχαμε για το σημαντικό αυτό θέμα. Επίσης χαιρετίζω το ψήφισμά σας και τις ερωτήσεις που υποβάλλετε για τις ανεξελίξεις διαπραγματεύσεις για την ανανεωμένη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών ε, της περιοχής Αφρικής, Καραϊβικής και ειρηνικού της χώρας ΑΚΕ. Οι διαπραγματεύσεις ε, προχωρούν με μέτριο ρυθμό. Ως επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας ε, οφείλω να είμαι ρεαλιστής. Όταν λήξει ε, στις 29 Φεβρουαρίου του 2020 η Συμφωνία Κοτονού δεν θα έχουμε προχωρήσει πολύ στις διαπραγματεύσεις. Οπότε θα χρειαστούν μεταβατικά μέτρα για το ενδιάμεσο διάστημα. Χαίρομαι που το Συμβούλιο α, υιοθέτησε μια απόφαση υπέρ της παράτασης της Συμφωνίας Κοτονού μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2020. Έτσι θα έχουμε μια πάγια νομική βάση που θα παραμείνει ενισχύ και κατά τη μεταβατική περίοδο. Η Επιτροπή Πρέσβεων Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΚΕ θα λάβει την τελική απόφαση μέχρι τα τέλη του Ιανουαρίου του 2020 το αργότερο. Σε αυτό το προηγμένο στάδιο των διαπραγματεύσεων, χαίρομαι ιδιαίτερος που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, διατρανώνει και πάλι τα βασικά στοιχεία που περιείχε και, τα τα προηγούμενα δύο ψηφίσματα, το 2016 και το 2018 το ευρωπαϊκό Κοινοβουλίου. Ε, εισακούγεται η άποψή σας. Έχετε ένα κυρίως αίτημα, την ενίσχυση της κοινοβουλευτικής διάστασης. Ε, ακόμη και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΚΕ. Πιστεύω, αγαπητέ Ευρωβουλευτέ, ότι ο ρόλος των ε, κοινοβουλίων θα πρέπει να ενισχυθεί στην ε, μελλοντική συμφωνία με τις χώρες ΑΚΕ. Βέβαια, με βάση και τις κατευθυντήριες διαπραγματευτικές γραμμές του Συμβουλίου, θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να γίνει στο επίπεδο των περιφερειακών πρωτοκόλων και όχι τόσο στο, σε επίπεδο βασικής ε, συμφωνίας ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΚΕ. Παρ' αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό της ενίσχυσης κοινοβουλευτικής διάστασης. Επίσης θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι οι συστάσεις της Επιτροπής προς το Συμβούλιο ε, το Δεκέμβριο του 2017 περιλάμβαναν και την πρόταση τα οι τρεις περιφερειακές κοινοβουλευτικές ε, συνελεύσεις να συγχωνευτούν σε μία ε, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Τελικά αυτή η πρόταση δεν συμπεριληφθήκε στις ε, διαπραγματευτικές οδηγίες του Συμβουλίου. Επίσης, χαιρετίζω την πρότασή σας για πολιτικό διάλογο. Μάλιστα, έχουμε υποβάλει προτάσεις στου ε, συνομιλητέ μας για σφαιρικό διάλογο που θα καλύπτει όλους του στόχου τη στόχους, και του τομεί πολιτικής. Επίσης, ε, συμμερίζομαι την ανησυχία σας για μια γνήσια πολυμερή εταιρική σχέση. Η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ξεκάθαρη επιδιώκουμε μία δέσμευση όλων των συμβαλωμένων μερών να διευκολύνουν την ενεργό συμμετοχή ε, μεγάλου φάσματος φορέων ε, σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Και σε ό,τι αφορά το αίτημά σα για ενίσχυση των διατάξεων για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή έμφυλης ταυτότητας ε, και την διαφύλαξη των δικαιωμάτων σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, θα ήθελα να σας πω ότι εστερνιζόμαστε τα, ε, τις απόψεις σας και έχουμε συγκεκριμένη γραμμή. Μέχρι στιγμής όμως οι προτάσεις μας ε, δεν έχουν τύχει θερμής υποδοχής ε, από πλευράς χωρών και οπότε θα συνεχιστούν αυτές οι διαπραγματεύσεις. Μέχρι στιγμής στην παράγραφο αυτή τα σχετικά σημεία έχουν μπει σε παρέθεση. Σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ιδιαίτερω τον προβληματισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και χώρε ΑΚΕ συνεχίζουν τι διαπραγματεύσει για ένα ισορροπημένο κείμενο που θα αναζητεί μια σημαντική συμβαστική λύση που θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα και των δύο μερών. Σε ό,τι αφορά τι συμφωνίε οικονομική εταιρική σχέση, θα ήθελα να σα υπενθυμίσω ότι είναι αυτόνομες διεθνείς σχέσεις, ε, συμφωνίες. Βέβαια, η συμφωνία ε, που θα ακολουθήσει την ε, Συμφωνία Κοτονού θα αποτελέσει ένα συμπαγές πλαίσιο για συνεργασία με τις χώρες ΑΚΕ και θα συνδέει όλες τις τωρινές και μελλοντικέ συμφωνίες οικονομικές εταιρικής σχέσεις που θα πρέπει να σέβονται βασικά και απαραίτητα στοιχεία. Τέλος, ό,τι αφορά την ερώτησή σας για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Ευπρόσδεκτη η ερώτηση και μου δίνει την ευκαιρία να ε, επαναλάβω ότι το θεματολόγιο του 2030 των ΗΕ Εθνών θα διαμορφώσει και τη μελλοντική μας εταιρική σχέση με τις χώρες ΑΚΕ. Ο σφαιρικός μας διάλογος με τις χώρες ΑΚΕ και η πολυμερής προσέγγιση θα χρειαστούν για να θεσπιστούν οι προϋποθέσεις και οι μηχανισμοί για την τακτική παρακολούθηση και εφαρμογή των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Εκ μέρους τώρα του ΕΛΚ, το λόγο έχει ο κύριος Γιώργη Χολβαϊνή για τρία λεπτά. Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα σε όλους, ε, καλό βράδυ σε όλους. Η συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών ΑΚΕ είναι αναπόφευκτη για να μπορέσουν να βρεθούν λύσει στα ζητήματα όπω η μετανάστευση, η αντιμετώπιση τη κλιματική αλλαγή, η πρόσβαση στην εκπαίδευση αλλά και τα ζητήματα ασφάλεια. Η συμφωνία του Κοτονού, η οποία είναι ακόμα ενισχύ, μα παρέχει ένα καλό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών. Η ενδεχόμενη καθυστέρηση τη θέση σε ισχύ ε, της νέας συμφωνίας ε, θα οδηγήσει σε προβλήματα για την Ευρωπαϊκή, την, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα βρεθεί σε μειονεκτική θέση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει ε, να ενισχύσει τα στοιχεία εκείνα τα οποία κρατούν τους ανθρώπους στις χώρες τους και που εξασφαλίζει την ασφάλεια. Το πιο βασικό στοιχείο της συνεργασίας αυτής είναι η μάθηση και η επαγγελματική κατάρτιση. Θέλω να αναφερθώ σε κάτι πολύ σημαντικό. Όταν μιλάμε για τις χώρες ΑΚΕ, η συνεργασία με θρησκευτικές οργανώσεις είναι αναπόφευκτη. Όμως αυτή τη στιγμή δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ε, στην υποσαχάρια Αφρική η περίθαλψη, η εκπαίδευση ε, κατά 50% είναι κάτι που το παρέχουν θρησκευτικές οργανώσεις. Μεταξύ λοιπόν οργανώσεων ε, ανάπτυξης θα υπάρχουν και οργανώσεις θρησκευτικέ. Στη νέα συμφωνία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να βρει μια λύση για να μπορέσει να διαχειριστεί το θέμα της μετανάστευσης ή τουλάχιστον να κάνει μια απόπειρα να επιλύσει τα μεταναστευτικά προβλήματα. Όπως ε, μόλις είπε και ο Υπουργός, ε, θα πρέπει να επικεντρωθούμε στους λόγους, στις αιτίες της μετανάστευσης και να βρούμε λύσεις έτσι ώστε οι άνθρωποι αυτοί να επιστρέψουν στη χώρα τους, σε μια χώρα όμως που θα, όπου θα υπάρχει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση, όπου θα υπάρχει ε, απασχόληση, θα επιτρέψει στους ανθρώπους αυτούς να ζήσουν τη ζωή τους με αξιοπρέπεια. Από το 2021 θα πρέπει να εφαρμοστούν ε, τα NDC και τα NDICI και θα μπορούσε να συμπεριληφθεί εδώ και το NDF ως ε, βασικός πόρος. Θα πρέπει να δούμε πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να συνδέσει τη Συμφωνία του Κοτονού και την οικονομική εταιρική σχέση. Αναμένουμε λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φτάσει σε μια συμφωνία που θα βοηθάει τους ανθρώπους να μείνουν στις χώρες τους και να μην μεταναστεύουν. Και επίσης ε, να ενισχύσουμε τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πλαίσια της συνεργασίας με τις χώρες ΑΚΕ. Ευχαριστώ εκ μέρους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το λόγο έχει ο κύριος Κάρλος Ζοχίνιο. Για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Η συζήτηση που γίνεται με πρωτοβουλία τη Επιτροπή Ανάπτυξη για τι ανεξελίξει διαπραγματεύσει για τη νέα συμφωνία εταιρική σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και χωρών ΑΚΕ είναι πολύ σκόπιμη ε, και χαιρετίζω τον Πρόεδρο για την πρωτοβουλία του. Θα πρέπει λοιπόν να συγκεκριμενοποιήσουμε με αποφασιστικότητα και ταχύτητα τους μηχανισμούς ε, αυτής της νέας συμφωνίας ε, που ανταποκρίνεται και σε γεωστρατηγικούς στόχους. Και μάλιστα την περασμένη εβδομάδα στο Κιγάλι της Ρουάντα είχαμε την 38η Κοινοβουλευτική Συνέλευση εις εκπροσώπηση, στην οποία συμπροέδρευσα ως επικεφαλής αντιπροσωπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στη συνεδρίαση λοιπόν εκείνη, οι ευρωβουλευτές που εκπροσωπούν περίπου πάνω από 100 χώρες και περίπου 2 δισεκατομμύρια ανθρώπους κατέληξαν σε σημαντική συνένεση να τηρηθούν και τα χρονοδιαγράμματα και οι εντολές ώστε να μπορέσουμε να οριστικοποιήσουμε τη συμφωνία μέχρι τον Αύριο του 2020 και να σφυριλατήσουμε μια κρατέα και σχέση μεταξύ ισοτήμων που θα εμπνέεται από το θεματολόγιο του 2030 και ε, θα στηρίζεται σε μια ε, σε ένα ελαστικό όραμα και προσέγγιση που θα συνδυάζει ε, τα οικονομικά και εμπορικά συμφέροντα με, τα, ε, με τους κοινούς στόχους της ε, βιώσιμης ανάπτυξης. Επίσης θα πρέπει να ενισχύσουμε και να εξορθολογήσουμε την κοινοβουλευτική διάσταση της συμφωνίας που είναι ειδοποιώς διαφορά σε αυτή τη γεωπολιτική ανταγωνιστική κατάσταση που επικρατεί. Έχω επίγνωση ότι το να μιλούμε για τη συμφωνία του Κοτονού δεν λέει και πολλά στους Ευρωπαίους πολίτες. Αν του εξηγήσουμε όμω πόσο σημαντικό είναι αυτό για να καταπολεμήσουμε την, την ερημοποίηση, τι ε, τις κλιματικές αλλαγές, τις αναγκαστικές μετακινήσεις, και τις συγκρούσεις λόγω ενδημικής φτώχειας ε, ε, και επίσης πόσο σημαντικό είναι να συγκεκριμενοποιήσουμε μια καλή συμφωνία με τις χώρες αυτές που θα είναι επωφελής για όλους, τότε θα πείσουμε και τους Ευρωπαίους ε, ότι είναι σημαντική αυτή η συμφωνία. Επίσης θα ήθελα να χαιρετήσω και να συγχαρώ τον Επίτροπο Μίμητσα για το εξαιρετικό έργο που έχει επιτελέσει. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Εκ μέρους της ομάδας Renew Europe το λόγο έχει η κυρία Χρυσούλα Ζαχαροπούλου. Για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Ε, όλοι γνωρίζουμε σε αυτή την αίθουσα ότι είναι συνδεδεμένη η μοίρα μας με αυτή τον χωρό και θα είναι ακόμα περισσότερο συνδεδεμένη στο μέλλον. Μόνο από κοινού μπορούμε να δώσουμε απαντήσεις ε, στις παγκόσμιες προκλήσεις, ξεκινώντας βεβαίως από τη διαχείριση της κλιματικής κρίσης την κρίση της βιοπικιλότητας. Οι φίλοι μας των χωρών ΑΚΕ κρούν τον κόσμο, τον κόσμο του κινδύνου, διότι οι επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών βάζουν σε κίνδυνο την επιβίωσή τους. Οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές είναι απαραίτητες ε, για να δράσουμε πριν είναι πολύ αργά. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε και επίσης το θέμα του ε, λαθρεμπορίου ε, άγριων ζώων αποτελεί μέρος ε, της προσπάθειας προστασίας της βιοπικιλότητας. Υπάρχει επίσης το θέμα των νέων και των γυναικών, ιδιαίτερα στην Αφρική. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρε ΑΚΕ πρέπει να δημιουργήσουν γέφυρε μεταξύ των νεολαίων του, στον τομέα τη εκπαίδευση, στον τομέα τη επιχειρηματικότητα, στον τομέα των ακαδημαϊκών, τον πολιτιστικό. Έτσι θα μπορέσουν να χτίσουν από κοινού το μέλλον του. Αλλά υπάρχει και το θέμα τη όρτα μεταξύ των δύο φύλων. Ε, η εκπαίδευση των γυναικών και η αναπαραγωγική και σεξουαλική εκπαίδευσή του. Είναι πολύ σημαντικό αυτό οι δυνατότητε των γυναικών να μπορέσουν να απελευθερωθούν. Είναι η καλύτερη, η καλύτερη, το καλύτερο στίχημα, η καλύτερη επένδυση για το μέλλον. Μετά από τόσα χρόνια εταιρική σχέση και ενώ υπάρχουν πλέον νέοι δράστε στα πλαίσια τη οικονομική συνεργασία, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί ε, να κάνει χωρί του ιστορικού τη συμμάχου. Είδαμε ότι οι χώρε ΑΚΕ θέλουν μια πραγματική εταιρική σχέση. Ε, εγώ όμω ω Ευρωπαία θέλω αυτή την πραγματική εταιρική σχέση. Έχουμε τα πάντα στα χέρια μα για να δημιουργήσουμε μια νέα σχέση που θα βασίζεται όλο και περισσότερο στη συνεργασία και στην αμοιβαία, στον αμοιβαίο σεβασμό. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστούμε. Εκ μέρου των Πρασίνων και άλλε, το λόγο έχει η κυρία Πιερέτ Χέρτσπεργκερ Φοφάνα. Δύο Για δύο λεπτά. Η νέα συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΚΕ θα είναι η ευκαιρία να δημιουργήσουμε θέσεις εταιρικής, σχέσεις, σχέσεις εταιρικές ε, σε ένα πνεύμα ισότητας, μια πραγματική εταιρική σχέση που δεν θα είναι πατερναλιστική. Όλα θα εξαρτηθούν από τα των διαπραγματεύσεων που είναι ήδη όμως προβληματικές. Ήδη με το ξεκίνημα, με το άνοιγμα στο ελεύθερο εμπόριο, πολλές χώρες ΑΚΕ δεν είναι σε θέση να ανταγωνιστούν τα φτηνά προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αυτή τη στιγμή πλημμυρίζουν τις χώρες του ΣΑΕΛ στην Αφρική. Το παράδειγμα τη γάλα σε σκόνη που έρχεται από την Ευρώπη και που πωλείται στι αφρικανικέ αγορέ είναι χαρακτηριστικό. Και βεβαίω ε, δεν μπορεί να το ανταγωνιστεί αυτό το τοπικό γάλα. Είναι ένα θέμα επικαιρότητα που ανησυχεί και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι χώρε ΑΚΕ. Όμω θα πρέπει να φροντίσουμε τα χρήματα για την ανάπτυξη να μην σχετίζονται με τα δρακόντια, μέτρα για τη μεταναστευτική πολιτική της Ένωσης που έχει γίνει ένα εργαλείο ε, με, ε, με δίκο που είναι και γίνει δίκο μαχαίρι. Έχει αυξηθεί ε, έτσι η δύναμη των εθνικιστών που μιλούν για λήψη ασφάλειας. Θα πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε ε, να εξαλείψουμε την φτώχεια, να προωθήσουμε την εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση, να προωθήσουμε την, μόνη, την νόμιμη μετανάστευση καθώς και τη δυνατότητα επιστροφής στη χώρα προέλευσης με εθελοντική ε, επανένταξη, να φτάσουμε δηλαδή σε μια συμφωνία που να αποκρίνεται, να αποκρίνεται στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Δεν πρέπει η αναπτυξιακή βοήθεια ε, να, να συνδυάζεται με πολύ υψηλά εμπόδια σε επίπεδο μετανάστευσης, ασφάλειας και περιβάλλοντος. Μια τέτοια πολιτική είναι ενάντια στις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις αρχές που θα πρέπει να διέπουν τις σχέσεις μεταξύ εταίρων. Το να επιβάλλουμε τέτοιες πολιτικές στις χώρες ΑΚΕ ε, μοιάζει πολύ με μια νεοαπικιακή πολιτική. Πρέπει ε, να μοιραστούμε με τους φίλους μας της χρόνια και τις σκέψεις μας, την ευφυΐα μας και να φτάσουμε σε μια συμφωνία που να προκρίνει τις προσδοκίες και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του χρόνο και. Ευχαριστώ. Εκ μέρους ομάδας Ταυτότητα και Δημοκρατία το λόγο έχει η κυρία Ντομίνικ Μπίλντ. Για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. στιγμή που από την Κίνα μέχρι τη Ρωσία όλοι έχουν αντιληφθεί το δυναμικό της Αφρικής, που θα είναι ήπειρο του 21ου αιώνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσεγγίζει τι διαπραγματεύσει αυτέ από δύναμη θέση και κατάσταση. Όχι μόνο γιατί τίποτα δεν κάνει για να διορθώσει, αντισταθμίσει την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, που είναι σημαντικό συνεισφορέα και πραγματικό παράγοντα, αλλά ουσιαστικά γίνεται, διαπιστώνει την αποτυχία του κοτονού. Γιατί ούτε ο πολυμερή διάλογο που εσαρκώθηκε από του θεσμού ε, δεν κατάφερε να φέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα, ούτε οι υποχρεωτικοί μηχανισμοί στέφθηκαν και με επιτυχία. Αποτυχία και στη μετανάστευση. Γιατί ενώ το άρθρο 13 ήταν αναποτελεσματικό, τελικά ε, εξαρτήσαμε όλη τη βοήθεια στον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών από τις χώρες προέλευσης, κάτι που θα έπρεπε ε, να ήταν ε, από τις πρώτες μας απαιτήσει. Επίσης, σε οικονομικό επίπεδο είχαμε πολύ χαμηλό, πενιχρό απολογισμό για το σύμφωνο της Αφρικής με πρωτοβουλία της Γερμανίας ήταν μια τρύπα μέσα στο νερό σε ό,τι αφορά την κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων. Το ίδιο θα ισχύσει και για το Γενικό Σχέδιο Δράσης που με στον φόδι τρόπο χαρακτηρίστηκε το σχέδιο Marshall για την Αφρική πώς ε, ήταν δυνατόν να έχουμε κάτι διαφορετικό όταν δεν συντρέχουν οι στοιχειώδεις προϋποθέσεις και οι στοιχειώδεις εγγύσεις. Είχαμε επίσης το τραγικό θάνατο 13 συμπατριωτών, γιατί απέναντι στην Ισλαμική τρομοκρατία οι Γάλλοι στρατιώτες δίνουν μόνοι τους τη μάχη. Και ενώ ε, οι διεθνείς δεσμεύσεις δεν τηρήθηκαν επί τότου, ε, το τίμημα που πληρώνουμε είναι με το αίμα μας. Ευχαριστώ. Εκ μέρους των Πρασίνων... Ε, συγγνώμη, εκ μέρους της GUE NGL. Το λόγο έχει ο κύριος ε, Μιγέλ Ουρμπάν Κρέσπο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πριν από ένα χρόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τι διαπραγματεύσει για τη σύναψη νέα συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και των 78, χρόνο των 78 χωρών ΑΚΕ. Οι διαπραγματεύσει αυτέ ε, περιλάμβανε στο αρχικό κείμενο την αντιμετώπιση προκλήσεων όπως η κλιματική αλλαγή και έδινε πιο πρωταγωνιστικό ρόλο στην κοινωνία των πολιτών και ενίσχυε τον κοινοβουλευτικό έλεγχο της συμφωνίας. Πριν από ένα μήνα όμως η Επιτροπή Ανάπτυξης ε, απέριψε σε μεγάλο βαθμό ε, το κείμενο αυτό και το ΕΛΚ ε, τώρα απειλεί να αλλοιώσει τη συμφωνία. Τι ζητάει το ΕΛΚ και η ακροδεξιά, το είχαν διατρανώσει και στην προηγούμενη του παρέμβαση. Είπαν ότι θέλουν να εξαρτήσουν την αναπτυξιακή βοήθεια από τον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών, που σε πολλές περιπτώσεις ισοδυναμεί με συστηματική παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είδαμε πολλές βαναυσότητες τα τελευταία χρόνια με τη χρήση των αναπτυξιακών κονδύλιων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, και την κακή του διαχείριση. Και τώρα θέλουμε να εξαρτούμε την αναπτυξιακή βοήθεια από τον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών. Αυτό κυρίε και κύριοι όχι μόνο είναι επέσχυντο και νεοαπικιακό, αλλά θα πρέπει να διατρανώσουμε ότι παραβιάζει όλα τα διεθνή πρωτόκολλα μια τέτοια συμπεριφορά. Ας μην διαπράξουμε λοιπόν αυτό το λάθος αύριο, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα πρέπει να ταχθούμε υπέρ μιας αναπτυξιακής πολιτικής που δεν θα υπηρετεί την Ευρώπη φρούριο, που δεν θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα της ακροδεξιάς, αλλά θα υπηρετεί τα, τους λαούς και τον πλανήτη. Από την αυριανή ψήφο μας θα εξαρτηθεί ποιους εξυπηρετούμε, τον κόσμο ή τους σκάβουμε το λάκκο το, του κόσμου. Εσείς θα αποφασίσετε. Σας ευχαριστώ. Το λόγο ο κύριος Άλβαρο Αμάρο για τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι πολύ σκόπιμη η διεξαγωγή αυτή τη συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο για αυτή την συμφωνία εταιρική σχέση μετά το κοτονού με τι χώρε ΑΚΕ. Ξεκινήσαμε μαζί αυτό το δρόμο με τους εταίρους από τις χώρες ΑΚΕ το 1975. Επίσης, η συμφωνία αυτή έχει τρεις θεμελιώδεις στόχους. Εξάλληψη της φτώχειας, μακροπρόθεσμα, βιώσιμη ανάπτυξη και συμβουλή, συμβολή στην συμπερίληψη των χωρών και στη παγκόσμια οικονομία. Θα πρέπει λοιπόν και η συμφωνία μετά το Κοτονού να εξυπηρετεί του ίδιου στόχου. Αυτό λέει και η διαπραγματευτική εντολή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η συμφωνία θα πρέπει να ενισχύσει τι θεμελιώδει αρχέ και ε, προσεγγίσει τη προηγούμενη έκθεση που ολοκληρώνεται τον επόμενο Φεβρουάριο. Θα πρέπει λοιπόν να υιοθετήσουμε συγκεκριμένα μέτρα και να προωθήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, να ενισχύσουμε τη δημοκρατία, την οικονομική ανάπτυξη και τι επενδύσει, ώστε να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή, να προωθήσουμε την ειρήνη και την ασφάλεια, να ε, συμβάλλουμε ε, στην εξάλληψη της φτώχειας και να τηρήσουμε τους ε, στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτά θα πρέπει να είναι η πηξίδα μας και για την νέα συμφωνία. Θα ήθελα επίση να κάνω τρία σχόλια για τι ενεξελίξει διαπραγματεύσει, γιατί σε πολλά με κάλυψαν οι συνάδελφοι. Θα πρέπει καταρχήν να διασφαλίσουμε και να διατηρήσουμε την κοινοβουλευτική συνέλευση στην επόμενη εταιρική σχέση Ευρωπαϊκή Ένωση ΑΚΕ. Και το αυριανό ψήφισμα αυτό ε, αναδεικνύει την ανάγκη ενίσχυσης της κοινοβουλευτικής συνέλευσης. Επίσης, το μελλοντικό θεσμικό ε, σχέδιο και πλαίσιο θα πρέπει να περιλαμβάνει μια κοινοβουλευτική συνέλευση εις εκπροσώπησης Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΚΕ. Σε χαίρο τον ε, Κάρλος Σορίνιο που συμπροέδρευσε στην ε, συνεδρίαση του Κιγκάλι και στην κοινή διακήρυξη αυτό ακριβώς αναφέρεται, η ενίσχυση της κοινοβουλευτική διάστασης. Και αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο σημείο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κόκκινη γραμμή μας στη μελλοντική συμφωνία. Επίσης, η πολυμέρεια είναι ο μοναδικό αποτελεσματικός δρόμο για μια υφόρο ειρήνη, οικονομική ευημερία και βιώσιμη ανάπτυξη. Μόνο έτσι θα καταφέρουμε να υλοποιήσουμε τους φιλόδοξους στόχους των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης στα διάφορα παγκόσμια φόρα. Και επίσης η εταιρική, η μας σχέση θα είναι σημαντικό πλαίσιο για τις κοινέ μας προτάσεις. Θα πρέπει να προωθήσουμε τις αρχές και τα ιδεώδη μας ε, για να μην μείνουν απομονωμένοι, γιατί όπως είπε και ο ποιητής, μπορεί ο καθένας μόνος του να πάει πιο γρήγορα, αλλά μαζί θα φτάσουμε πιο μακριά. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε ιδιαίτερη έφαση στην πολυμέρεια, σε επίπεδο κοινοβουλευτικό, σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και σε επίπεδο δημόσιας διοίκησης. Και επίσης, θα ήθελα να προσθέσω, θα πρέπει να εμπλέξουμε πιο ενεργά την κοινωνία των πολιτών στην πολιτική διαδικασία. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε τους στόχους μας και να έχουμε και πολλά, πολλές εκδηλώσει στην οποία θα αναδεικνύουμε την ε, συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και θα προσπίσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Μόνικα Σιλβάνα Γκονσάλες. Για ένα λεπτό. Απουσιάζει. Οπότε η κυρία Μονίκα Σεμέντο. Για ένα λεπτό επίσης. Και η κυρία Μόνικα Σεμέντο από ό,τι φαίνεται απουσιάζει ή όχι. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την προηγούμενη εβδομάδα είχα την ε, τιμή να παραστώ στην 38η Μεικτή Κοινοβουλευτική Συνέλευση με τις χώρες Ακέστο και Κιγκάλι στη Ρουάντα με τους ε, συναδέλφους μου εκεί που εξέφρασαν την λύπη τους για το ότι οι διαπραγματεύσεις ε, για μετά το Κοτονού καθυστερούν περισσότερο από όσο περίμεναμε, αλλά συμφωνήσαμε ότι οι ε, δυνατότητες αυτών των χωρών ε, κυρίως ε, οφείλονται στην νεολαία, την οποία πρέπει να προωθήσουμε τώρα. Θα πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε τον δυναμικό αυτών των ανθρώπων. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι έχουν εμπλακεί στις διαβουλεύσεις οι οργανώσεις της νεολαίας. Αν ναι, σε ποιο επίπεδο και αν όχι, δεδομένου του ότι οι διαπραγματεύσεις ε, συνεχίζονται ακόμα, θα περιληφθούν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Στρίκα έχει τον λόγο τώρα για τους πράσινους. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, βρισκόμαστε σε μία στιγμή κέρια. Η νέα συνθήκη αυτή θα δώσει νέα ορμή σε μια ισχυρή συνεργασία και χαιρόμαστε που ακούμε ότι πλησιάζουμε στην τελική φάση σύναψης μιας συμφωνίας. Όμως υπάρχουν ακόμα κάποια προβληματικά ζητήματα που επικεντρώνονται στο ζήτημα της μετανάστευσης και της κινητικότητας. Γι' αυτό εστιάζω σε αυτό. Η συνθήκη βασίζεται στην αρχή της ισότητας και της κοινή ευθύνη. Αλλά αν δείτε την πρόταση κειμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει πολύ συγκεκριμένες απαιτήσεις για τις χώρες ΑΚΕ, όπως επανειστοχή, ενίσχυση συνοριακών ε, ελέγχων, καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης, ενώ σε αντάλλαγμα δεν έχει καμία δέσμευση η Ευρωπαϊκή Ένωση για την νόμιμη μετανάστευση. Έτσι οι χώρες αυτές δεν θα μπορούν να έχουν τα εμβάσματα χωρίς ε, κάποια εναλλακτική για την μετανάστευση εργασίας. Ε, δεν πρόκειται για μια ισότητα. Όσον αφορά την κοινή ευθύνη, θεωρώ πως η μόνη διάταξη για τους πρόσφυγες και τη διεθνή προστασία είναι πολύ ε, χλωμή. Η Αφρική φιλοξενεί πολύ περισσότερους πρόσφυγες από εμάς. Γιατί δεν υπάρχει μια σοβαρή δέσμευση για την υποδοχή των προσφύγων, είτε μέσω χρημάτων, είτε μέσω της επανεγκατάστασης. Έτσι θα μοιραζόμασταν την ευθύνη. Επίσης, θα ήταν και σύμφωνο με το Παγκόσμιο σύμφωνο του ΟΗΕ και βεβαίως ε, θα έχουμε περισσότερους πρόσφυγες εάν κολλήσουν στις χώρες διέλευσης χωρίς πρόσβαση σε άσυλο. Οπότε, εάν η παράγραφος αυτή είναι ακόμα στην διαπραγμάτευση, φροντίστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει κάτι και για την μετανάστευση, την κινητικότητα και την διεθνή προστασία. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Ζωάου Φεχέιρα για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Οι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών ΑΚΕ, των χωρών δηλαδή Αφρικής, Καραβικής και Ειρηνικού, θα πρέπει να είναι μια γνήσια συνεργασία και εταιρική σχέση για την ανάπτυξη. Χωρίς νεοπικικές πρακτικές και με σεβασμό της κυριαρχίας αυτών των χωρών. Το μελλοντικό πλαίσιο συνεργασία θα πρέπει να αναγνωρίσει και να διαφυλάσει την ακαιρεότητα και την ενότητα των χωρών ΑΚΕ. Απορρίπτουμε λοιπόν τις προσπάθειες του Διέρη και Βασίλευε. Η... Να επιβάλλουμε πάση θυσία ε, εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Ένωση τη Συμφωνία Οικονομική Εταιρική Σχέση παρά τη βούληση των χωρών ΑΚΕ, προσπαθώντα να τι διχάσουμε στα πλαίσια των μελλοντικών μα διαπραγματεύσεων. Θα πρέπει να μην ε, ε, ε, ενισχύσουμε την υποτέλεια, αλλά την ανεξαρτησία των χωρών ΑΚΕ. Και γι' αυτό θα πρέπει να στηρίξουμε τα παραγωγικά του συστήματα ε, και την αυτονομία και τη συνοχή τους. Θα πρέπει να προωθήσουμε την ανάπτυξη δημοσίων υπηρεσιών στην υγεία, στην παιδεία, στην εξυγίαση του ίδιου και στην επεξεργασία αποβλήτων. Θα πρέπει να αξιοποιηθεί το χώριο δυναμικό της κάθε χώρας. Επίσης, να ενισχύσουμε το ρόλο του Ευρωπαϊκού Αναπτυξιακού Ταμείου με παρά με κονδύλια που θα χρηματοδοτούν τέτοιες προτεραιότητες. Επίσης θα πρέπει να προσέξουμε τις πολιτικές μας και να μην εξαρτήσουμε την αναπτυξιακή βοήθεια από, την τήρηση όρων για τη μετανάστευση. Δεν θα πρέπει να εξάγουμε νεοφιλελεύθερα νεαπικιακά μοντέλα που απέδειξαν ότι είναι καταστροφικά. Επίσης, θα πρέπει το χρέος του αναπτυσσόμενων χωρών να το διαγράψουμε. Αυτό είναι απαραίτητη χειρονομία δικαιοσύνης και κάτι ε, που ε, εγκρίθηκε στην πρόσφατη ε, συνέλευση του Κιγκάλη θα πρέπει να ενισχυθεί η κοινοβουλευτική διάσταση και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό το λόγο κύριος Πιέτρο Μπαρτόλο. Κυρία Πρόεδρε, είπαν ακόμα πάρα πολλέ οι ανοιχτές ε, ε, στα θέματα τα οποία είναι υπό διαπραγματεύση. Η βιώσιμη ανάπτυξη, η μειώσιμη τη φτώχεια, ε, η στάθμη των δικαιωμάτων, η κατάσταση της δημοκρατίας, η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και η κλιματική αλλαγή. Αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία θα μα οδηγήσουν σε μια κοινή ενισχυμένη συνεργασία μετά το 2020. Η Συμφωνία του Κοτονού μας οδήγησε βεβαίως στον διάλογο και τη συνεργασία και είχαμε σημαντικές επιτυχίες. Αλλά ας είμαστε ειλικρινείς, ακόμα απέχουμε πάρα πολύ από τους στόχους της μείωσης, της φτώχειας και της ένταξης των χωρών αυτών στην παγκόσμια οικονομία. Οπότε θα πρέπει να συνεχίσουμε στην πορεία του ανοιχτού κοινοβουλευτικού διαλόγου και να μην ε, ξεχνάμε ποτέ τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις δημοκρατικές αρχές, το κράτος δικαίου που πρέπει να αποτελέσουν βάση της συνεργασίας μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαρή Πιέρ Βεντρέν έχει τον λόγο. Ευχαριστώ κυρία Αντιπρόεδρε. Κύριε Πίτροπε, το μέλλον των σχέσεών μα μετά το Φεβρουάριο του 2020, δηλαδή και ολοκλήρωση τη Συμφωνία του Κοτσονού, το διαγωνισμό του Τεκμνέ, ήταν στο κέντρο των συζητήσεων μα την περασμένη εβδομάδα στο Κιγκάλι. Ω αντιπρόεδρος τη Κοινοβουλευτική επιτροπή Ευρωπαϊκή Ένωση ΑΚΕ, λυπάμαι που αυτό το πολυμερέ πλαίσιο, στο για το οποίο δεσμευόμαστε όλοι εδώ, απειλείται από αυτές τις διαπραγματεύσεις. Ε, μια πραγματική εταιρική σχέση, όπου έχουμε όλοι να κερδίσουμε, ε, θα υπάρξει μόνο εφόσον ενισχυθεί η κοινοβουλευτική διάσταση. Είναι αλήθεια ότι η λειτουργία αυτή της ε, συνέλευση πρέπει να μεταρρυθμιστεί για να είναι πιο αποτελεσματική, αλλά δεν μπορούμε ε, να την καταργήσουμε. Προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κράτο δικαίου, ε, στόχοι βιώσιμη ανάπτυξη, αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, Αυτέ Εκεί, αυτές, εκεί θα βρούμε λύσεις για τα ζητήματα αυτά μόνο να δράσουμε από κοινού. Και η διπλωματική, κοινοβουλευτική διπλωματία μάλλον πραγματικά ε, δημιουργεί ε, βήματα πρόοδου. Φτάσαμε σε μια κοινή προσέγγιση για την COP25 στη Μαδρίτη σε λίγε μέρε. Θέλω να στήσω για άλλη μια φορά την, Ευρωπαϊκή, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Συμφωνία των Παρισίων είναι ένα κεντρικό στοιχείο αυτή τη μελλοντική εταιρική σχέση. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Εβίνιν Τσίρ για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να τονίσω ε, κάποια σημαντικά πράγματα και απευθύνομαι προς την Κομισιόν και προς τα κράτη-μέλη. Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι στόχοι βίωσιμη ανάπτυξης της χιλιετίας, ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι θεμελιώδει ελευθερίες, το κράτος δικαίου, η δημοκρατία. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά για να στηρίξει η συμφωνία αυτή και την κοινωνία των πολιτών. Η ποικιλομορφία στην κοινωνία επίσης είναι πάρα πολύ σημαντική. Γιατί ο δημοκρατικός χώρος ε, μικραίνει συνεχώς παγκοσμίω για τις